Le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εστονίας, πρόεδρος Ήλβες. Liebe Kolleginnen und Kollegen, αγαπητοί Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να εξαιρετική μου χαρά να χαιρετίζω τον κύριο Τόμας Ήλβες στο Κοινοβούλιο. Επέστρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς ήταν επί σειρά ετών Ευρωβουλευτής. Σήμερα έρχεται δεύτερη φορά ως πρόεδρος της Εστονίας. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ε, καλωσορίζω και σας δίνω και αμέσως τον λόγο. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της Εστονίας. Κυρίες και κύριοι, ζητώ συγγνώμη, η φωνή μου είναι βραχνιασμένη. Κάτι κόλλησα στην Εστονία. Πριν από 10 χρόνια έφυγα από αυτή την αίθουσα για να πάω